για την ανάπτυξη δορυφορική τεχνολογία για να διαταχθούν επικρατά ζητήματα παγκόσμια παρακολούθηση πτήσεων. Τελεία. Αυτό είναι ο τίτλο. Ο κύριος Κράμερ πρώτος. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Κυρία Επίτροπε, αξιότιμη συνάδελφη, κυρία Πρόεδρε. Εξ ονόματο τη Επιτροπή Μεταφορών θα ήθελα να καταθέσω προφορική ερώτηση με θέμα ανάπτυξη δορυφορική τεχνολογία για να καταστούν εφικτά τα συστήματα παγκόσμια ε, παρακολούθηση πτήσεων. Πάρα πολλές τραγωδίε έδειξαν ε, μερινού συστήματος. Υπάρχει ανάγκη για ε, μια ακριβή και μόνιμη ε, αναγνώριση και τοπισμό των αεροσκαφών. Θυμάστε τις τραγικές ιστορίες της 370 της Malaysian Airlines και της Air France 447 και πολλές ακόμα πτήσει. Ε, θα μπορούσε κανείς να θυμηθεί. Μόλις 30% ε, του παγκόσμιου εναερίου χώρου ε, καλύπτεται σήμερα και παρακολουθείται. Αυτό εμποδίζει και την έρευνα και τη διάσωση. Χρειάζεται λοιπόν οπωσδήποτε να δράσουμε. Και μία από τις πολλά υποσχόμενες δυνατότητες είναι η παγκόσμια παρακολούθηση με τη δορυφορική τεχνολογία. Με αυτόματη ε, αυτό επιτρέπει και καλύτερο έλεγχο και καλύτερη διαχείριση της και κυκλοφορίας, αλλά πάνω απ' όλα περισσότερη ασφάλεια και περισσότερη αποτελεσματικότητα και έλεγχο και λιγότερο κόστος για τις υποδομές. Δηλαδή ε, είναι τριπλό το όφελος. Η Επιτροπή μας είναι πεπισμένη ότι οι κανόνες θα πρέπει να επαναξεταστούν έτσι ώστε να σώζονται ανθρώπινες ζωές. Και η Διεθνή Ένωση ε, Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας, η ΚΑΟ, συμφωνεί. Δηλαδή και η Επιτροπή μας και ο Διεθνής Οργανισμός παρακαλούν τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών, ITU, ε, στην παγκόσμια διάσκεψη που θα γίνει στη Γενέβη τον Νοέμβριο, να ε, προβεί στην απαραίτητη καταχώρηση συχνοτήτων ραδιοφάσματος. Είναι σαφή τα ερωτήματά μας. Ποια είναι η γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο αφορά την τεχνολογία παγκόσμιας δορυφορικής παρακολούθησης πτήσεων, ποια είναι η θέση της Επιτροπής εν ώψη της παγκόσμιας διάσκεψης να δώσει τις αναγκαίες συχνότητες ραδιοφάσματος για την υποστήριξη τέτοιων συστημάτων. Περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον την απάντησή σας κυρία Επίτροπε και σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Και σας ευχαριστούμε που θέσατε την ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Επίτροπε, έχετε λόγο για να απαντήσετε. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, ε, θα σας ε, μιλήσω για τέταρτη φορά για ένα θέμα το ίδιο σημαντικό με τα υπόλοιπα. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η τεχνολογία που είναι δορυφορική και αφορά τις πτήσεις και είναι μια θετική εξέλιξη διότι κατόπιν αυτών των τραγωδιών της ε, πτήσης 447 France τον ε, Ιούνιο του 2009 ξεκινήσαμε με το εντατικό αυτό έργο τόσο ώστε να μπορούμε να παρακολουθήσουμε τι γίνεται με τα αεροπλάνα και να μπορούμε να εντοπίσουμε που είναι τα αεροσκάφη που έχουν κάποιο πρόβλημα. Επίσης είχαμε και την τραγωδία της πτήσης 370 ε, της Malaysia Airlines του Μάρτιο Μάρτιο του 2014, οπότε και τότε ενδιαν μας και τον Ιούλιο του 2015 μα ζήτησαν ε, να μπορέσουμε να γνωμοδοτήσουμε ε, όσον αφορά την πρόταση αυτή για τον ε, κανονισμό 965 του 2012 και να δούμε τι θα γίνει με αυτές τις συσκευές εντοπισμού και τα συστήματα παρακολούθησης και με έρευνα και με νομοθεσία προχωρούμε και έχουμε ως μπούσουλα την απόδοση. Θέλουμε να βρούμε κάποιες εμπορικές, τεχνολογικές λύσεις και θέλουμε τις τεχνολογίες που να χρησιμοποιούν οι πάροχοι που να είναι κατάλληλο για τον σκοπό που χρησιμοποιείται. Και νομίζουμε ότι με τους νέους κανόνες θα έχουμε την κατάλληλη ευελιξία για να μπορέσουμε να καλύψουμε κάποιες τεχνικές επιλογές που ισχύουν και για σήμερα αλλά και για το μέλλον όπως το Γκαλιλαίο ε, έρευνα και διάσωση και το ε, EDS. Επίσης με αυτούς τους κανόνες έχουμε μαζί μας τα κρατη και έχουμε τρεις αρχές. Ε, ότι δηλαδή πρώτα-πρώτα θα πρέπει να υπάρχει τεχνολογική ουδετερότητα και θα πρέπει ε, να βασίζεται η λειτουργία πάνω στην απόδοση και να υπάρχει κάποια αυτόματη μετάδοση των πληροφοριών από τα αεροσκάφη αυτό να γίνεται με ακρίβεια και να αφορά έρευνα, διάσωση και επίσης ε, την ερευνητική δραστηριότητα. Επίσης θα πρέπει να δούμε πώς ε, το σχετικό υλικό θα μπορεί να καταστήσει σαφές ότι δεν θα διαταράσει ε, τη παρακολούθηση της πτήσης. Όλα αυτά ε, σε σχέση και με την τραγωδία της πτήσης της Malaysia Airlines. Οπότε είπαμε, οι αεροπορικές εταιρείες αλλά ε, και οι εταιρείε κατασκευή αεροπλάνων θα πρέπει να βρουν τι πιο αποτελεσματικέ προ λύσει και ήδη έχουμε υποβάλει την πρόταση αυτή του ε, νομοθετήματο στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Οπότε θα πρέπει πριν τα τέλη του έτου να έχει υιοθετηθεί το σχετικό νομοθέτημα και η ΚΑΟ, ο Οργανισμό Πολιτική Αεροπορία, επίση θέλει να προσαρμόσει όλους τους δικούς του κανόνες ανάλογα με αυτές τις προσπάθειες και έτσι να υπάρχει ίντερνετ που για τους ε, επιβάτες τέτοιες λύσεις μέσω της δορυφορικής τεχνολογίας και έτσι να υπάρχει καλύτερη ε, επικοινωνία αέρα εδάφους οπότε έτσι ε, να μπορούμε να παρακολουθήσουμε από εδάφους την πορεία της πτήσης τώρα πάλι για τις προσπάθειες τεχνολογίας θέλουμε εμείς να τονίσουμε ότι αυτή είναι μία πιθανή λύση γιατί υπάρχουν και άλλες. Υπάρχουν διαφορετικές επιλογές οι οποίες έχουν ε, περιγραφεί ε, σε μια τεχνική έκθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτή η έκθεση υποβλήθηκε στην ΙΚΑΟ. Οπότε είπαμε ότι θα κάνουμε αυτή την διάσκεψη των ράδιο ε, τηλεπικοινωνιών τέλο πάντων και με συμμετοχή της Διεθνής Ένωσης Τηλεπικοινωνιών ITU ήδη για αυτή τη διάσκεψη των επικοινωνιών έχει ε, αποφασίσει το Συμβούλιο και ελπίζουμε ότι θα προχωρήσουμε με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου και συνεργασία με τα κράτη-μέλη θα προχωρήσουμε σε αυτή τη ε, διάσκεψη επικοινωνιών και θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσει. Εν κατακλείδη, εμεί θέλουμε να υπάρχει ε, ADS-B, δηλαδή αυτή η εξαρτημένη επιχείρηση, σε σχέση με τον κανονισμό της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνίων ITU. Επίσης, θέλουμε να ετοιμάσουμε αυτήν την διάσκεψη επικοινωνιών και τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να δώσουν το πράσινο φως όσον αφορά το, την δορυφορική εξαρτημένη επιτήρηση εκπομπή ADS-B και αυτά τα μηνύματα ε, και η παρακολούθηση να γίνει σύμφωνα με τα πρότυπα του Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας, ΚΑΟ. Αυτά και σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος, κυρία Επίτροπε. Και τώρα, να ακούσουμε τις απόψεις των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Μαρινέσκου πρώτος, για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, ε, δυστυχώς θα πρέπει ε, να σας πω ότι είναι ε, τραγικά αυτά τα ε, συμβάντα και που ζήσαμε τελευταία και δεν υπάρχει κανένα καλό σύστημα παρακολούθησης των πτήσεων. Όπως είπαμε, μόλις 30% του εναέριου χώρου μπορεί να παρακολουθείται συνεχώς. Μεγάλα τμήματα του εναρίου χώρου πάνω από την Αφρική δεν παρακολουθούνται γιατί δεν υπάρχει η υποδομή εκεί και η τεχνολογία. Το σημερινό σύστημα είναι πολύ ακριβό και πολύ αναποτελεσματικό. Δεν μπορούν να εντοπίζονται σε πραγματικό χρόνο όλες οι πτήσεις και δεν γίνεται ε, καλή χρήση του εναρίου χώρου. Υπάρχει όμως η τεχνολογία, υπάρχει η τεχνική λύση για να εξασφαλίζεται μια καλή κάλυψη. Είναι το ε, ADSB και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ε, είναι δορυφορική αυτόματη εξαρτημένη επιτήρηση και εκπομπή. Αυτό που χρειάζεται είναι να δοθεί ε, συχνότητα στο ραδιοφάσμα Μπορεί να γίνει αυτό στο πλαίσιο λοιπόν της Παγκόσμιας Διάσκεψης Ραδιοεπικοινωνιών του 2015, WRC 15, το Νοέμβριο. Η επόμενη αντίστοιχη διάσκεψη θα γίνει μετά από τέσσερα χρόνια. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για να μην χάσουμε άλλη μία τέτρα αιτία. Ε, θα είναι πολύ αποτελεσματικό το σύστημα αυτό για τις δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης αλλά και τις πτήσει πάνω από τους ωκεανούς, κυρίως τις υπερατλαντικές. Υποστηρίζουμε αυτή την ε, θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την καλωσορίζουμε. Ξέρουμε ότι και ο ΙΚΑΟ είναι στο πλευρό μας. Παρακαλώ να κάνετε ό,τι χρειάζεται να γίνει πραγματικότητα αυτό στην λόγω διάσκεψη. Ευχαριστώ, η Πρόεδρος. Και τώρα και σας ευχαριστώ που τηρήσατε και το χρόνο σας κύριε Μαρινέσκου. Ακολουθεί η κυρία Άντερσον από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αριθμιστικά σώματα έχουν δεχτεί ότι πρέπει η παρακολούθηση των πτήσεων με δορυφόρο να γενικευτεί. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία δορυφόρων είναι έτοιμη αλλά βέβαια υπάρχει το θέμα των συχνοτήτων και το θέμα δεν αφορά μόνο διασώσεις αλλά και την αύξηση της δυνατότητας να βοηθούνται αεροσκάφη ώστε να μολύνουν λιγότερο το περιβάλλον και να ακολουθούν ασφαλέστερες διαδρόμους. Πρέπει λοιπόν να γίνουν όλα αυτά. Οι ταξιδιώτες και οι οικογένειές τους πρέπει να θυσυχαστούν. Και γι' αυτό παρακαλώ τους συναδέλφους στην Ολομέλεια να υποστηρίξουν το ψήφισμα σας κατευχαριστώ. Ε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Η κυρία Φώστερ τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. ευχαριστώ Επιτροπή. Δέχομαι το ερώτημα του συναδέλφου μας Μιχαήλ Κράμερ. Είναι κατάλληλη η στιγμή. Είναι ηρωνικό ότι εγώ το θέμα το έχω θέσει πριν από δεκα, πάνω από 13 χρόνια όταν ήμουν στην Επιτροπή Βιομηχανίας. Εκείνη την εποχή υπήρχε η μεγάλη αύξηση των κινητών και βρισκόμασταν πριν το Γαλιλαίο. Τι έκανε λοιπόν η τεχνολογία, προόδευσε ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση ώστε να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τέτοια συστήματα παρακολούθησης των πτήσεων. Το κοινό ενδιαφέρεται επίσης για να διαλευκάνονται καλύτερα, πιο εύκολα τα δυστυχήματα παραδείγματος χάρη, έτσι ώστε να χορηγήσουμε τα εργαλεία για να γίνει αυτό, να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Χαίρομαι λοιπόν για αυτή τη συζήτηση και φυσικά θα στηρίξουμε τον εισηγητή και όσο μας. Ευχαριστούμε ο κ. Στέλιτσκα. Είναι προφανές ότι όχι μόνο υποστηρίζουμε την ερώτηση, το θέμα, αλλά έχουμε συμβάλει και στη σύνταξή του. Νομίζω ότι σήμερα φάνηκε ότι η Κομισιόν κάνει ό,τι μπορεί και αυτό το εκτιμεί ιδιαίτερα η ομάδα μου. Δεύτερον, μας επιβεβαιώσατε ότι οι δέσμοι για την αεροπορία, για την αεροπλοεία θα συμπεριλαμβάνει και αυτή την πρόταση και εξετάζοντας τώρα τα τρία βασικά στοιχεία θα έλεγα ότι το backup supply δεν αφισβητείται πια από κανέναν όσο για την τεχνολογική ουδετερότητα θα έλεγα ναι μεν αλλά θα κοιτάξουμε και την αξιολόγηση. Το κύριο θέμα είναι να υπάρχουν συνδυασμένες μεταφορές, να υπάρχει δυνατότητα συνδυασμού. Μπορεί να μην είναι το φτηνότερο η φτηνότερη μέθοδος αλλά είναι η καταλληλότερη. Και τέλος για την ε, κανονικότητα. Για το γενικό φάσμα δεν έχω τίποτα να πω. Κύριε Σερτούγκ, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Επίτροπε, προφανώς υποστηρίζω και εγώ την πρόταση του συναδέλφου Κράμε. Αυτή τη φορά θέλω να αφιέρω στο χρόνο αγόρευσής μου στη γενική αεροπλοεία και την επιχειρηματική. General and Business Aviation. Αυτό το σύστημα θα πρέπει να επεκταθεί και στα μικρά αεροσκάφη. Ε, ε, Γαλλικός Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας έχει υπολογίσει ότι κατά μέσο όρο έχουν ετησίω 15 δυστυχήματα και στις μισές περιπτώσεις είναι και θανατηφόρα. Εδώ πραγματικά υπάρχει έδαφος για περισσότερα δυστυχήματα που θα πρέπει και μπορούμε να αποτρέψουμε. Γι' αυτό ζητώ να έχουμε ε, την συνολική εισαγωγή του συστήματος ATSB και κατά τα το 2008 ήδη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε εκπονήσει έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας ε, που απαιτούσε κάτι τέτοιο και μέχρι τώρα συγεί ηχθείως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας εκλυπαρώ να δραστηριοποιηθείτε και εσείς κυρία Επιτροπέ, στην Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Και τώρα ακολουθεί η διαδικασία ΚΑΤΣΙΑΙ. Σας ευχαριστώ, κυρία Επίτροπε, κυρία Πρόεδρε. Ασφάλεια πάει να πει σύστημα ανείχνευσης και εντοπισμού των αεροπλάνων που έχουν κάποιο πρόβλημα. Θα πρέπει να μπορούμε να τα καλύψουμε. Τώρα καλύπτουμε μόνο 30% του παγκοσμίου εναερίου χώρου. Υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι όπου δεν υπάρχει καμία εποπτεία, ας πούμε, στους ωκεανούς ή πάνω από τα δάση. Οπότε είπαμε ότι τώρα θέλουμε με το σύστημα ADS-B να έχουμε καλύτερη διαχείριση της εναερίας κυκλοφορίας. Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε τι προβλήματα έχει η ασφάλεια, τι πρόβλημα μπορεί να έχει το καινούργιο σύστημα και οπότε υπάρχει τώρα ένα χρονοδιάγραμμα ούτως ώστε να τεθεί σε λειτουργία στην Ευρωπαϊκό Εναεριοχώρο το σύστημα ADS-B. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε. Κύριος Μαριάς, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι αεροπορικές τραγωδίες στην Ευρώπη φέρνουν στη μνήμη μας άσχημες αναμνήσεις και την απώλεια εκατοντάδων συνανθρώπων μας. Οι αιτίε των αεροπορικών δυστυχημάτων μένουν σχεδόν πάντα ανεξιχνίαστες και χωρίς κανείς να γνωρίζει τα αίτια των αεροπορικών αυτών δυστυχημάτων. Σήμερα που βρισκόμαστε στην εποχή της ψηφιακής εποχής και των τεχνολογιών, είναι απαράδεκτο μόνο το 30% των αεροπορικών εταιριών να παρέχουν συστήματα εντοπισμού πτήσης. η τεχνολογία αυτή θα βοηθήσει τις κυβερνήσεις τους παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας και τις αεροπορικές εταιρείες να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας ενώ παράλληλα θα αυξηθεί σημαντικά η ασφάλεια των αερομεταφορών. η επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει άμεσα μέτρα για να χρησιμοποιείται παγκόσμια το υποσυζήτηση σύστημα φροντίζοντας παράλληλα να μην παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να υπάρχει σεβασμός στα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν είμαστε πάρα πολλοί παρόντες. Δεν ξέρω αν θέλει κανένας άλλος λόγο. Σας παρακαλώ κάντε λίγη ησυχία να ακούσουμε την Επίτροπο να μας απαντήσει και να μπορούμε να την ακούμε. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτέ, η Επιτροπή θα ήθελα να ευχαριστήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και τον κύριο Κράμερ για αυτή την προφορική ερώτηση, η οποία αντικατοπτρίζει συγκεκριμένου προβληματισμού και προσδοκίε των Ευρωπαίων πολιτών. Εμεί είμαστε ολόθερμα υπέρ του να γίνουν ε, βήματα προόδου όσον αφορά την παρακολούθηση των αεροσκαφών όπω το ADSB και να γίνουν επίση και άλλα βήματα προόδου όσον αφορά την νομοθεσία αυτά τα οποία σα είπα στην εισήγησή μου. Ελπίζω ότι έτσι ξεκαθαρίζεται πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πασχίζει να υπάρξει ένα κοινό σύστημα ασφαλές και ε, να είναι κάποια λύση αποτελεσματική και από πλευράς κόστος όσον αφορά την παρακολούθηση ε, των, των αεροπλάνων. Οπότε θα πρέπει να δούμε κατά πόσον με το Συμβούλιο θα μπορέσουμε έγκυρα να έχουμε εγκρίνει τη συγκεκριμένη νομοθεσία. Και σας ευχαριστώ η πρόεδρος. Εμείς σας ευχαριστούμε κυρία Επίτροπε για την ε, τόσο σύντομη περιεκτική σας απάντηση. Εδώ κλείνει αυτή η συζήτηση. Έχουμε επομένω την πρόταση ψηφίσματο και θα γίνει ψηφοφορία σήμερα για αυτό το θέμα. Ακόμα υπάρχει χρόνο μέχρι τι 11 και 30. Οπότε θα διακόψουμε μέχρι τότε τη συνεδρίαση για να ετοιμαστείτε για την ψηφοφορία.